Του κατάλογους θα του βρείτε στα πρακτικά τη συνεδρίασης και αν μέχρι την των ε, πρακτικών δεν έχω ακούσει σχετική αντίρρηση θεωρώ ότι θα εγκριθούν αυτοί οι διορισμοί αυτέ οι αλλαγέ.